Συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε. Παρακαλώ την τον εισηγητή να έρθει στο Προεδρία. Η κυρία Μορβάη έχει ένα διαδικαστικό. Ναι, κυρία Πρόεδρε, έχω διαδικαστικό. Μήπως θα πρέπει να ακυρώσουμε αυτή την ε, ακρόαση και την Ερευνητική Επιτροπή ε, λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος, ε, έλλειψη των Ευρωβουλευτών, γιατί άμα γυρίσει η ε, κάμερα πάρει μία λήψη της ε, αίθουσας, τη βλέπουμε άδεια έδρανα. Ενώ όταν είχαμε τη ρέκτη στα για την Ουγγαρία ήταν κατάμεστη αίθουσα. Έχουμε ανθρώπους που ρεψοκινδυνεύουν τη ζωή τους για να καταγγείλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε μόνο 10% των ευρωβουλευτών που δίνουν το παρόν και δείχνουν ενδιαφέρον. Επίσης δεν πρόκειται να πάμε με την αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον και να συμμετέχω σε εργασίες. Μα κυρία Μορβάη δεν είναι δικαστικό αυτό. Συμφωνώ μαζί σας ότι η κοινή αίθουσα, η απουσία πολλών συναδέλφων είναι αξιολύπητη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε λίγοι δεν έχουμε δικαίωμα να θέτουμε ερωτήσει. Άλλωστε, η συνεδρίαση αυτή αναμεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι ελάχιστε ευκαιρίε έχουν να παρουσιάσουν την κατάσταση στο φως της δημοσιότητας. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας και τον εισηγητή μας και να σας δώσω λίγες εξηγήσεις για την οργάνωση της απογευματινής συνεδρίασης. Έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δυσαρεστηθούν μερικοί. Ε, σκοτώστε με. Έτσι είχαμε αποφασίσει, αλλά θα αναλάβω την ευθύνη ως πρόεδρος, γιατί βλέποντας και την αίθουσα, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις αλλαγές. Μόνο ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές ε, θα θέσουν ερωτήσεις. Και χαίρομαι, κυρία Μορβάη, που προσωπείτε τους ε, μη εγγεγραμμένους, γιατί στη μόνη παρούσα από τους μη εγγεγραμμένους, οπότε θα λάβετε και στο λόγο, αλλά μόνο ο εισηγητής, οι σκιώδεις εισηγητές κυρία Μορβάη θα θέσουν ερωτήσεις και έχουν ένα δίλεπτο το πολύ. Και θα είμαι πραγματικά πολύ αυστηρή και θα χρησιμοποιήσω και το σφυρί στην, ε, στο χρόνο μιλιές, Θα το πολύ ε, δύο λεπτά λοιπόν και μία συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό. Δύο μάλλον ερωτήσεις δύο λεπτών συν ε, δύο συμπληρωματικές το πολύ, δηλαδή έξι λεπτό καθένας για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη σε εγκαίρος. Βέβαια, άμα μας περισσέψει χρόνος, μπορώ να δώσω το λόγο και σε άλλους. Εννοείται. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ καλή αυτή η ρύθμιση, αλλά μόνο έτσι θα έχουμε καλή συζήτηση. Γιατί την περασμένη φορά είχαμε τόσες πολλές ερωτήσεις που δεν προλάβαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Καλωσορίζω θερμά τον κύριο Χέρτ Standard που είναι εκπρόσωπο της Belgacom και ο κύριος Λίμπαρτ, Γενικός διευθυντή της Belgacom. Και επίσης ε, για το δεύτερο γύρο ερωτήσεων να καλωσορίσω τον κύριο Φρανκ Ρόμπεν, που είναι ο Βέλγος Επόπτη Προστασία Δεδομένων και είναι συνεισηγητή για την υπόθεση Belgacom. Λυπούμε που δεν μπορώ να καλωσορίσω και τον κύριο Λόμπαν, είναι η πολιτική της καινής έδρας που ασκεί ο κύριος ε, Σεριάν Λόμπεν. Γιατί στο παρελθόν και εκπρόσωποι της Αμερικανικής κυβέρνησης και της Ολλανδικής ε, ακολούθησαν την ίδια πολιτική. Είναι πραγματικά αξιολύπητο που δεν έρχονται εκπρόσωποι των κυβερνήσεων να λογοδοτήσουν μπροστά στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στους κυρίους Στάνταρτ και Λίμπερτ για σύντομες εισαγωγές και μετά θα περάσουμε σε γύρω ερωταπαντήσεων. Ο κύριος Στάνταρτ πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, στις 16 Σεπτεμβρίου η Belgacom επισήμανε ότι στα πλαίσια της ε, αποκατάστασης ασφάλειας ε, των ε, δικτύων πληροφορικής διαπίστωσε ότι έγινε θύμα δικτυοπαραβίασης με τις αποκαλύψεις αυτές ε, σχολιάστηκε το θέμα ευρέως και στον Βελγικό και στο Διεθνή Τύπο. Εκ μέρους του Βελγακόμ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην ακρόαση αυτή και να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση των διαφόρων ε, περιστατικών πριν απαντήσω στις απορίες σας. Έτσι θέλω να συμβάλλουμε επικοδομητικά ελπίζω στην συζήτηση που έχετε στην Επιτροπή σας. Καταρχήν να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στις 21 Ιουλίου του 2013 οι εμπειρογνώμονες της BelgaCom έκρουσαν το κόδωνα του κινδύνου ασφάλειας διαπιστώνοντας κάποιες ανομαλίες στο εσωτερικό δίκτυο της BelgaCom, εξαιτίας ενός κακόβουλου λογισμικού. Οπότε καλέσαμε την εταιρεία Fox IT που μαζί με τους εμπειρογνώμονες της Belgacom έκαναν εμβριθεί έρευνα των ανομαλιών. Στις 12 Ιουλίου διαπιστώσαμε δικτυοπαραβίαση με τη χρησιμοποίηση ενός πολύ περίπλοκου και άγνωστο για το σύστημα της Belgacom EU. Στις 19 Ιουλίου υποβάλλαμε μήνυση κατά γνώστου στην ε, εισαγγελία των Βρυξελών. Άρχισαν αμέσω ε, έρευνες ε, από την εισαγγελία με την Ειδική Υπηρεσία Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, τη Στρατική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Ασφάλειας του Βελγίου. Μάλιστα, ε, συνεχίσαμε και εμείς ταυτόχρονα τις εσωτερικές μας έρευνες, ενώ συνεργαστήκαμε και με τις δημόσιες αρχές. Προσπαθήσαμε πρώτα να ε, αναγνωρίσουμε τον ιό αυτό και να δούμε τι ε, κακό προκάλεσε και αν χρησιμοποιήθηκαν και δεδομένα των πελατών μας. Τελικά βρήκαμε τον ιό αυτό μόνο στο εσωτερικό δίκτυο πληροφορικής της Belgacom και όχι στα δίκτυα κινητής ε, ή σταθερής ε, τηλεφωνίας της Belgacom. Τα... Επίσης ε, δεν επηρεάστηκε η τράπεζα δεδομένων των πελατών μας. Αυτή έμεινε άθικτη. Παρακολουθήσαμε εκ του της Δραστηριότητε αυτού του ιού και ταυτόχρονα σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες και τις αρμόδιες αρχές προσπαθήσαμε να χαράξουμε στρατηγική και να αντιμετωπίσουμε τις ζημίες αυτού του κακόβουλου λογισμικού. Και μάλιστα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να καταστρέψουμε διαρθρωτικά τον ιό αυτό. Και μαζί με την εταιρεία Fox IT καταφέραμε να εκπονήσουμε κάποια εργαλεία για την εκαθάριση του συστήματος. Από τη στιγμή που εφαρμόσαμε επιτυχώς ε, αυτά τα θέματα και τελικά ολοκληρώσαμε στις 14 με 15 Σεπτεμβρίου τις διαδικασίες εκαθάρισης. Έχουμε 26.600 ε, συστήματα πληροφορικής στο σύστημα της Belgacom και 124 από αυτά είχαν μολυνθεί από τον ιό. Αυτά τα μολυσμένα συστήματα είτε αντικαταστάθηκαν είτε απομονώθηκαν αμέσως. Έγινε με ιδιαίτερα προσοχή όλη αυτή η διαδικασία γιατί ήταν ιδιαίτερα τεχνική και έπρεπε να ακολουθηθεί συγκεκριμένη σειρά στις διάφορες αυτές επιχειρήσεις. Πάντως έχει γίνει η εκαθάριση του συστήματος χωρίς να έχουμε αντίκτυπο, αρνητικές επιπτώσεις στο υπόλοιπο δίκτυο στους πελάτες. Τελικά συνεχίζουμε να ελέγχουμε εξονυχιστικά όλο το σύστημα για να αποφύγουμε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό. Έκτοτε όμως, μετά την ε, ε, αποκατάσταση της ασφάλειας του συστήματος, δεν έχουμε βρει άλλες ενδείξεις ε, δικτυοπαραβίασης ή υποκλοπής. Και ευελπιστώ ότι με την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας θα διαλευκανθεί το θέμα και θα βρεθούν οι αυτούργοι και τα κίνητρά τους. Προς το παρόν δεν έχουμε αντικειμενικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε τις ε, οικοτολογίες ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε τίποτα. Επίσης δεν μπορούμε να σας ε, δώσουμε πληροφορίες που εμπίπτουν στο δικαστικό απόρριτο. Γιατί συνεχίζεται η δικαστική έρευνα από την Βελγική Εισαγγελία και δεδομένης της ποινική διαδικασία δεν μπορούμε να σας κοινοποιήσουμε πληροφορίες που θα διακυβεύσουν την πορεία της ε, συζήτησης, ούτε να σας δώσουμε πληροφορίες που θα διακυβεύσουν την ασφάλεια του δικτύου πληροφορικής της Belgacom. Αυτή τη διευκρίνηση θα κάνω πριν ε, δηλώσω την προθυμία μου να απαντήσω στις απορίες σας. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάντερτς. Ο κύριος Λίμπαρτς, ο Γενικός Γραμματέας της Belgacom έχει το λόγο. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω, λέει ο κύριος Λίμπαρτς. Καλώς αυτό μας αφήνει χρόνο για τις ερωτήσεις. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Μωράης. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και τους δύο, λέει ο κύριος Μωράης. Να αναφερθώ στο νομικό κομμάτι. Είναι προφανές από αυτά τα οποία μας είπατε ε, και μεταφέρατε αυτά τα ευρήματα μετά την εσωτερική έρευνα στη Βελγική Εισαγγελία. Εμείς ε, ε, εξετάζουμε τους ισχυρισμούς του Σπίγκελ και θέλουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να μάθουμε όσο μπορούμε περισσότερα για το πόσο έχει υπονομευθεί η οργάνωση της Belgacom και ψάχνουμε πληροφορίες γύρω από αυτό. Εκτιμούμε ότι δεν μπορείτε να πείτε πολλά για το νομικό κομμάτι, αλλά εφόσον εσείς έχετε προσφύγει στον Βελγό Ισαγγελέα σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η ποινική διαδικασία. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ε, ποια είναι απλά η προσπάθεια αυτή, η κυβερνοεπίθεση, hacking, και πόσο όλα αυτά έχουν σχέση με τους ισχυρισμούς του Σπίγκελ. Οι ισχυρισμοί του Σπίγκελ ήσαν αληθείς ή δεν ήσαν αληθείς. Δεύτερον, ο Βέλγος Πρωθυπουργό μίλησε για παραβίαση της ακαιρεότητας της δημόσιας επιχείρησης. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σοβαρό το συμβάν αυτό για την ακαιρεότητα της επιχείρησής σας και πού ακριβώς τοποθετείτε ε, την κατάσταση σήμερα. Έχουμε μπροστά μας την προσπάθεια να καταλάβουμε τα αισθήματά σας, να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Belgacom. Είναι μια μεγάλη ακέραια βελγική επιχείρηση, αλλά εξυπηρετεί και τα βελγικά όργανα και ε, σε ποιο βαθμό υπονομεύθηκε η επιχείρησή σας στα πλαίσια της προσφοράς υπηρεσιών προς το Βέλγιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, ε, θα είμαι αυστηρή, από την επόμενη ερώτησή σας θα έχετε λιγότερο χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να δώσω μια απάντηση γύρω από τα θέματα που έχουν σχέση με τη δικαστική έρευνα. Στο Βέλγιο, όταν μια επιχείρηση στον κλάδο της, ε, της, των τηλεπικοινωνιών ε, διαπιστώσει ε, κυβερνοπειρατεία είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει τις πληροφορίες στις δικαστικές αρχές. Το κάναμε αμέσως μόλις διαπιστώσαμε ότι πράγματι υπήρξε μια οργανωμένη διείσδυση στο δίκτυό μας και στην ακαιρεότητα των πληροφορικών μας συστημάτων. Το ότι καταθέσαμε μήνυση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι γνωρίζουμε το ποιος είναι αυτός που έκανε την διείσδυση αυτή. Το άρθρο του Σπίγκελ είναι ένα από τα πιθανά σενάρια, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα αρχίσουμε να πιθανολογούμε. Το να εντοπισθούν οι ένοχοι είναι ε, δουλειά του εισαγγελέα, του ανακριτή ε, που θα ασχοληθεί με το θέμα. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα γύρω από αυτό σχετικά με τα ευρωπαϊκά όργανα και τις υπηρεσίες της Belgacom μέχρι σήμερα. Αυτό το λογισμικό δεν βρέθηκε παρά μόνο στα εσωτερικά συστήματα λειτουργίας και υπάρχουν πραγματικά μονοτικά σημεία ανάμεσα στα εσωτερικά μας συστήματα και στα εξωτερικά σταθερή συγκινητής τηλεφωνίας τα οποία δεν βρήκαμε κανένα τέτοιο κακόβουλο αν θέλετε δίκτυο. Δεν έχουν φυγεί ούτε οι υπηρεσίες προς τους πελάτες μας ούτε και τα δίκτυα δεδομένων μας. Το θέμα της διείσδυσης μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε και τοποθετήθηκε στη σωστή του διάσταση. Και αμέσως μετά εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε την υπογραφή ε, του συγκεκριμένου ιού και την διαδικτυακή διεύθυνση ε, του φορέα του συγκεκριμένου ιού μεταφέραμε τις πληροφορίες αυτές και στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία και στην Εισαγγελία και στα ευρωπαϊκά όργανα που ασχολούνται με την ασφάλεια του συνόλου των ευρωπαϊκών οργάνων. Είναι ενήμερες δηλαδή οι δικές σας υπηρεσίες ασφαλείας και έχουν τα στοιχεία τα οποία θα σας επιτρέψουν να ελέγξετε και να επαληθεύσετε το εάν έχετε θυγεί από κακόβουλους ιούς. Αλλά αν κρίνουμε από το τι συνέβη στα δικά μας συστήματα δεν έχει υπάρξει μεταφορά του malware, του κακόβουλου λογισμικού στα δικά σας δίκτυα. Βος δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση με, την, ε, με το τελευταίο σχόλιο σας απαντήσατε και στην ερώτηση που ήθελα να κάνω. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι και τεχνικός εμπειρογνώμων, αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πού εντοπίστηκαν τα δεδομένα, πού μεταβιβάστηκαν, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε το σημείο που έγινε η επίθεση και τι είδους δεδομένα ενδεχομένως ε, υποκλάπηκαν πιο το περιεχόμενό τους και επειδή υπάρχουν και υποψίες ότι ενδεχομένως η δίκτυο παραβίαση έγινε από την Μεγάλη Βρετανία, πώς καταλήξατε σε αυτή την υποψία ή ε, ήταν τα μέσα ενημέρωση αυτά που ανέφεραν τη Μεγάλη Βρετανία ως πηγή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λούμπερτ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν ήρθε κανείς σε εμά και ότι όσα γνωρίζουμε από όσα γνωρίζουμε δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας οδηγεί σε κάποιον συγκεκριμένο δράστη ή κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο. Έχετε κάποια παραπάνω ερώτηση? Μπορούμε δηλαδή να υποθέσουμε ότι θα μπορούσαν την επίθεση αυτή να την έχουν διεξάγει κάποια άλλα κράτη. Τουλάχιστον αυτό εικάζει κανείς από τα λεγόμενα της εφημερίδας. Και ε, στην ερώτησή μου σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων αυτών. Έχετε κάποιο στοιχείο βασισμένο στο οποίο να μπορείτε να μας πείτε αν έχουν παραβιαστεί ιδιωτικά, προσωπικά δεδομένα, εάν έχει γίνει κάποια υποκλοπή από αυτό το κακό βιολογισμικό. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε σε καμία περίπτωση διαπιστώσει αδίποτε ανομαλία στα δεδομένα του δικτύου ή στα δεδομένα τα οποία διαμετακομίζονται μέσω του δικτύου μας. Οι ανομαλίες διαπιστώθηκαν μόνο από την πλευρά της πληροφορικής εσωτερικών δικτύων της επιχείρησής μας οι ε, σερβερ Windows σαν παράδειγμα, ορισμένες εφαρμογές Office που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης, όχι όμως τα εξωτερικά δίκτυα. Σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση, η προέλευση αυτής της παραβίασης δεν γνωρίζουμε τίποτα, τίποτα που να μας φέρει κοντά στους δράστες, την ταυτότητα των δραστών, καμία απόδειξη ή ένδειξη Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα σε αντίθεση με την προηγούμενη ακρόαση θα μιλήσω και ως ως συγγήτρια. Θα θέσω την ερώτηση στα Ολλανδικά. Είπατε στην αρχή ότι η κυβερνοεπίθεση αυτή εντοπίστηκε από τους ειδικού της Belgacom. Είναι αλήθεια αυτό ή η επισήμανση έγινε από κάποιον άλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι δεν γνωρίζετε τους ε, αυτοργούς ούτε τα κίνητρά τους ή τι επιδίωκαν. Όταν όμως βλέπουμε πώς έδρασαν αυτοί οι hackers, βλέπουμε ότι έχουμε κάποια κοινά σημεία με την επίθεση του 2011. Και εκεί είχαμε παρεμβολές στα δίκτυα πληροφορικής. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε και στις δύο περιπτώσεις ε, ε, ε, προσπάθειες των μυστικών υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας. Μήπως αυτές ανορχίστρωσαν την επίθεση. Και τώρα πια έχει γίνει εξηγήση του δικτύου. Έχει αποκατασταθεί ασφάλεια. Και μια και... Ε, τι γίνεται με, τις, τους ρούτερ, τα μόντεμ της Cisco γιατί ακούστηκε ότι δεν έχει γίνει αποκατάσταση ασφάλειας. Επίσης, ε, ακούσαμε ότι θα γίνει μια μετεγκατάσταση της IMX προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, εκεί θα είναι πολύ πιο ευάλωτο το σύστημα στην πειρατεία των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Και μια πιθανολόγηση, μια θεωρητική ερώτηση. Έχετε καμία υποψία μήπως η τελευταία επίθεση σχετίζεται με αυτά που αναφέρονται για την επιχείρηση σοσιαλιστής ε, των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ε, οι δικέ μας υπηρεσίες ανακάλυψαν τον ιό και το κακόβουλο λογισμικό και συνεννοηθήκαμε αμέσω ε, με τη Microsoft και τη Hewlett Packard που είναι οι προμηθευτές μας. Διαπιστώσαμε ότι επρόκειται για ιό. Στην αρχή είδαμε την ανομαλία στο σύστημα. Δεν αντιληφθήκαμε αμέσω ότι πρόκειται για ιό. Διαπιστώσαμε τι ανομαλίε, καλέσαμε την ειδική ε, υπηρεσία Fox και εκείνοι μα είπαν ότι πρόκειται για ένα κακόβουλο λογισμικό, για ένα πολύ ε, εξεζητημένο ιό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το modus operandi, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Με βάση πληροφορίες που λάβαμε και που ε, διαβεβάσαμε ε, θα ήθελαμε να διαπιστώσουμε αν το modus operandi ήταν αντίστοιχο ή παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε το 2011 κατά των κυβερνοεπιθέσεων στις κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε ολοκληρώσει την εκαθάριση, την εξηγίαση όλων των συστημάτων και την αποκατάσταση της ασφάλειας σε όλο το σύστημα πληροφορικής της Belgacom και συνεχίζουμε παρακολούθηση του συστήματος. Δεν βρήκαμε πάντως ίχνη ιού. Και, η και τα μόντεμ Cisco είναι πια καθαρά. Σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση IMX στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχω ιδέα. Ε, δεν μεταφέραμε εμεί το σύστημα IMX στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το πέρα συνεδρίασης θα σας δώσω σε ό,τι αφορά το κωδικό επιχείρηση σοσιαλιστής που ανέφερε το άρθρο του Σπίγκελ, θα ήθελα να τονίσω ότι το άρθρο του Σπίγκελ είναι ένα από τα πιθανά σενάρια. Δεν μπορούμε ούτε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το αποκλείσουμε. Ευχαριστώ. Ε, δεν ε, έχω άλλε ερωτήσει συμπληρωματικές. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά να πω ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπος από τις ε, βρετανικές ε, μυστικές υπηρεσίες και πιστεύω πως πρέπει να καλέσουμε όλες τις κυβερνήσεις των ε, κρατών μελών να αντιδράσουν άμεσα διότι πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με θέμα εθνικής ασφάλειας και την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη. Είναι μια επίθεση, εξωτερική επίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω πως πρέπει να επιμείνουμε στην συνέχιση των συζητήσεων. Τώρα, να σας ευχαριστήσω καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε εδώ. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με το εσωτερικό σύστημα ασφαλείας στα δίκτυα πληροφορικής σας. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς πώς επηρεάστηκαν τα συστήματα πληροφορικής στα οποία αναφερθήκατε. Τι ακριβώς παραβιάστηκε. Επίσης, ε, εκτός από τους δικούς σας σερβερς υπάρχουν άλλοι όπως οι BICS που παραβιάστηκαν εξωτερικοί ή άλλες δραστηριότητες με τις οποίες συνδέεστε που έπεσαν θύματα αυτής της επίθεσης. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζετε εάν η BICS προσφέρει και άλλες υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Από κύριε Στάντερ και Ίσως μπορώ εγώ να απαντήσω στην ερώτησή σας για, το, για την εταιρεία BICS που είναι θηγατρική της ε, Belgacom. Φροντίζουν για τις ε, καλές επικοινωνίες ανάμεσα στα διαφορά δίκτυα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει ότι οι servers της ε, BICS ασχολούνται με την περιαγωγή και κλείσαν και SMS. Όταν θέλουμε να συνδέσουμε εκατοντάδες παρόχους στον κόσμο, οι BICS ασχολούνται. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πάροχη. Είναι ένας πελάτης της BICS. Ε, η BICS ήταν ένα εσωτερικό τμήμα της Belgacom στο παρελθόν και αποσπάστηκε και ιατρική μόνο τον Αύγουστο του 2012. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή συνδέσεις ανάμεσα στο δίκτυο της ε, BICS και στο δίκτυο της Belgacom. Και πράγματι βρήκαμε κακόβουλο λογισμικό και στην Belgacom και στην BSES. E Τώρα να απαντήσω στη, σε μια ενδεχόμενη επόμενη ερώτησή σας για το αν πραγματικός ο στόχος ήταν η BICS. E Δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να εκφράσουμε κάποια άποψη γι' αυτό. Να προσθέσω επίσης ότι επίσης δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς έγινε αυτή η επίθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ένδειξη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό το malware βρισκόταν στο εσωτερικό σύστημα πληροφορικής και ανάμεσα σε αυτό και στα εσωτερικά μας δίκτυα. Και φυσικά ελέγξαμε τα δίκτυα δεν βρήκαμε τίποτα εκεί, κανένα malware στις εφαρμογές ε, του Office οι οποίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά στην ε, εταιρεία. Όπως είπα, έχουμε πάνω από 26.000 ε, συστήματα. Έχουμε τους servers με Windows, έχουμε τερματικά PC, όπου εκεί εντοπίστηκε αυτό το malware, σε 124 από αυτά. Και σε 60-70 υπολογιστές δηλαδή. Μία επόμενη ερώτηση, κάπως πιο γενική. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτή η επίθεση, αυτή η παράνομη δίσδυση στο σύστημα πληροφοριών σας προήλθε από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Θα λέγατε ότι αυτό θα επηρεάσει την επιχείρησή σας και θεωρείτε εσείς ότι είναι αποδεκτό η κυβέρνηση του Βελγίου να μην αντιδράσει σε αυτή την παραβίαση της επιχειρηματικής σας ακαιρεότητας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, είναι υποθετική αυτή η ερώτηση, όπως είπατε κι εσείς. Οπότε πρέπει να δώσω και μία πολύ προσεκτική απάντηση. Αλλά να σας παραπέμψω στη δήλωση του Πρωθυπουργού ο οποίος είπε ότι το περιστατικό αυτό ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε. Όμως ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχυρίζονται πως γνωρίζουν ποιος έκανε την επίθεση αυτή και να είστε σίγουρος ότι αν μάθουμε και εμείς θα δράσουμε. Μάλιστα. Περνάμε τώρα εφόσον λείπουν οι υπόλοιπε και στην κυρία Ένστα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, να πω ότι εδώ διακυβεύεται η ακαιρεότητα των ε, τηλεπικοινωνιών και των ε, υποδομών τηλεπικοινωνιών μιας ολόκληρης χώρας. Πρέπει να αντιληφθείτε τις διαστάσεις αυτού του θέματος δεν είναι μόνο τα δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται. Έχει χαθεί εδώ ένα κομμάτι της εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα εμάς. Και πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε μια διεξοδικότατη ανάλυση του συμβάντος και να μην σταθούμε στην επιφάνεια. Τώρα, όπως είπα, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Στο Spiegel αναφέρεται ένα QI, Quantum Insert, ένα εξειδικευμένο λογισμικό. Και ήθελα να ρωτήσω, εσείς τι γνωρίζετε γι' αυτό, τι είναι αυτό, είναι πρόγραμμα, είναι λογισμικό, ποιος το έφτιαξε, ποιος το δημιούργησε, τι πληροφορίες έχετε για αυτό το QI. Έπειτα, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη για αυτό που είπατε για το ποιοι επλήγησαν από την επίθεση. Είπατε ότι οι πελάτες δεν επλήγησαν και ότι η επίθεση έγινε μόνο στα εσωτερικά συστήματα πληροφορίας. Εντάξει, αλλά εγώ διάβασα ότι το 2010 ήδη συνέβη, έγινε αυτή η επίθεση, τώρα έχουμε 2013 και εγώ θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι ζημιές που έγιναν από αυτό, ποια είναι τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις. Και τέλος, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, μιλήσατε για ένα σχέδιο πρόληψης. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το σχέδιο πρόληψης. Εντάξει, μας είπατε ότι δεν είμαστε σίγουροι και ακόμα κάνουμε ελέγχου, αλλά μπορείτε να μας ενημερώσετε περισσότερο και ακριβέστερα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάντερ, κύριε Λίμπερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το λογισμικό, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Και σίγουρα όσοι το σχεδίασαν και το ανέπτυξαν ε, είχαν στη διάθεσή τους ε, πολλές ε, δυνατότητες τεχνικές και πολύ σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Άλλες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας δώσω παρά μόνο ότι ο ιός ήταν όντως πολύ εξεζητημένος και περίπλοκος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ημερομηνία του 2010 που αναφέρατε. Όντως, εμείς ανακαλύψαμε τον ιό στα τέλη Ιουνίου και αμέσως λάβαμε δράση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ημερομηνία της ε, παραβίασης, ε, Δύσκολο είναι να προσδιοριστεί η ακριβή ημερομηνία. Συνεχίζεται άλλωστε η έρευνα, η δικαστική έρευνα για το θέμα αυτό. Και σε ό,τι αφορά τη, τη στρατηγική πρόληψης, θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες γιατί μας δεσμεύει το απόρριτο. Δεν μπορούμε καν να σας αποκαλύψουμε τα μέτρα που λάβαμε μετά την επίθεση αυτή. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ποια είναι η γενική μας θέση. Μαζί με άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών έχουμε κάνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αυτά για την πρόληψη. Τα υπόλοιπα με δεσμεύει για τα υπόλοιπα το απόρριτο. Ναι, ε, όπως ε, ρώτησα, θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την ανάλυση που κάνατε. Εάν κάνετε κάποια ανάλυση σε αυτό το λογισμικό και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο πρόληψης. Πιστεύω πως έχετε περισσότερη ευθύνη από αυτή που ισχυρίζεστε. Πώς έχετε. Θα μπορούσα απλώ να σας πω ότι έχουμε αποκαταστήσει την ασφάλεια, έχουμε εξοντώσει τον ιό. Τώρα για τις διάβλους παρίσφρησης, διείσδησης Έχουμε εντατικοποιήσει την παρακολούθηση του δικτύου σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να γίνει πιο αδιάβλητο. Σε ό,τι αφορά τη δική μας στρατηγική, εμείς ως επιχείρηση τηλεπικοινωνιών χειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα και έχουμε καθήκον και υποχρέωση να μεριμνούμε διαρκώς για την ασφάλεια των δικτύων μας. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα και ίσως ε, έτσι μπορούμε να δούμε με διαφορετικό πρίσμα το περιστατικό αυτό. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα λοιπόν είναι ότι πρόκειται για δράστη που είχε στη διάθεσή του πολύ σημαντικούς πόρους και τεχνολογία εχμής. Και ακόμη και συστήματα πολύ προστατευμένα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τέτοια κυβέρνοεπίθεση. επίθεση. Από τη στιγμή που ο δράστης έχει τέτοια, τέτοιους στη διάθεσή του και τέτοια προηγμένη τεχνολογία, κανείς δεν μπορεί να μείνει αλόβητος ε, ή να το αντισταθεί. Το θέμα είναι πώς ε, μια επιχείρηση μπορεί να προστατεύσει το δίκτυό της. Αυτή είναι η ευθύνη μας και το μέλημά μας. Βέβαια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τις επιχειρήσεις μόνες τους να καλύψουν ε, τα δίκτυά τους θα πρέπει να υπάρχει γενική ρυθμίση για πρόληψη αλλά και για καταστολή σε περίπτωση παραβίασης. Μάλιστα πρόσφατα εγκρίνεται και σχετική οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Η οδηγία αυτή είναι ήδη ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να δούμε αν και σε τοπικό, εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεννόηση και να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στις δημόσιες αρχές, ίσως με συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών, ώστε να καταπολεμηθούν τέτοιου είδους παραβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα και εγώ στον τύπο και τις ε, επιθέσεις της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας εναντίον ε, κάποιων βελγικών συστημάτων, την SFR και τους πελάτες σας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λέτε εσείς ότι δεν είναι κάτι το σαφές το ότι η Βρετανή και η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας είναι υπεύθυνη προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει οι ποινικέ διαδικασίε έτσι ώστε να βρεθούν, να εντοπιστούν οι δράστε μέσω των ανακρίσεων και τη συλλογή στοιχείων. Πάντω ο στόχο του εγκλήματος συνήθω έχει μια ξεκάθαρη θέση. Ποια είναι η θέση σα, λοιπόν σαν θύμα, σαν Belgacom και σαν εκπρόσωπος επίσης των μεμονωμένων θυμάτων που είναι οι πελάτες σας. Ποια είναι η θέση σας για την ανακριτική διαδικασία και τι κινήσεις έχετε κάνει μέχρι τώρα έτσι ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. Και δεν φοβάστε ότι ο δικός σας ρόλος ως θύματος στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω και των ειδικών σας, των νομικών συμβούλων σας. Μήπως ρόλος σας λοιπόν είναι να βοηθήσετε και εσείς στον εντοπισμό της ταυτότητας των δραστών. Και η ερώτηση ε, είναι μια ερώτηση που έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι. Γιατί τα υπόλοιπα θύματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην εκπροσωπούνται από νομικούς συμβούλους ε, στηριζόμενους βέβαια και εδραζόμενους σε τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί τα δικαιώματα των θυμάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να προστατευθούν. Ευχαριστώ πολύ. Όταν λέτε ότι εμείς έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και έχουμε έναν σαφέστατο ρόλο ως θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό είναι σωστό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προσφέραμε την απόλυτη συνεργασία μας με τις, τις δικαστικές αρχές. Τώρα, ποια είναι τα δικαιώματά μας ως θύματα, αν θέλετε, σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, είμαστε αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν τη μήνυση. Έχουμε καταθέσει μήνυση εναντίον αγνώστων και αυτό μας δίδει κάποια δικαιώματα, όχι στην παρούσα ίσως φάση της ανάκρισης, αλλά στη συνέχεια. Εάν υπάρξει ε, ε, μια κατηγορία, αν απευθυνθεί μια κατηγορία, τότε σε αυτή την περίπτωση η Belgacom θα έχει άμεση πρόσβαση στον φάκελο τον ανακριτικό. Αυτή είναι η ποινική διαδικασία που εφαρμόζεται στο Βέλγιο. Αυτό θα είναι το δικαίωμά μας ακριβώς ως θύμα αυτής της επίθεσης. Κυρία Μόρβαϊ. Πιστεύετε ότι θα είστε ηθικά δεσμευμένοι και νομικά δεσμευμένοι για να χρησιμοποιήσετε όλα σας τα μέσα, όλους σας τους εμπειρογνώμονες και όλες τις διεθνείς σας συμμαχίες και εταιρικές συνεργασίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται στον τύπο δεν έχουν τον τελευταίο καιρό γίνει κάποια βήματα από πλευρά σας και αυτό ίσως κάποιος να εκπλήσει. Υποθέτω βέβαια ότι υπάρχει ένας εισαγγελέα ο οποίος εφαρμόζει τον νόμο, ο οποίος όμως δεν θα έχει και πάρα πολλές τεχνικές αρμοδιότητες, ενώ σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δηλαδή εσείς και οι εταίροι σας θα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο. Έχουμε την ηθική ευθύνη όπως είπατε και θα πρέπει ε, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες. Το ότι στην παρούσα φάση της ανάκρισης δεν έχουμε ακόμα πλήρη πρόσβαση ε, στην διαδικασία αυτό είναι σαφές. Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ανάκρισης θα έχουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε πάντως μέχρι τώρα είναι να συνεργαζόμεθα πλήρως με τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και οι εμπειρογνώμονες οι εσωτερικοί μας συνεργάζονται με, συνεργάζονται σε επίπεδο έρευνας πληροφορικής με την δικαστική αστυνομία στο Βέλγιο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. Και υποθέτουμε λοιπόν ότι για μας και ε, για τους πελάτες μας ε, είναι βασική προτεραιότητα το συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους θα ήθελα ίσως να μάθω αν όπως το λέγουν τα μέσα ενημέρωσης η υπεύθυνη της παροβίασης της ακεραιότητας των συστημάτων σας μπόρεσε να παρακολουθήσει τις τηλεφωνικές κλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε έχει δίκιο η κυρία Μορβάη, εμπλεκόμεθα πλήρως. Όχι, είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να λέγει ότι παρακολούθησαν τις τηλεφωνικές σας συνδιαλέξεις. Λοιπόν, έχουν ζητήσει πέντε συνάδελφοι, ένα και τριάντα για τον καθένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπάρξουν και απαντήσεις. Τρεις ερωτήσεις πρώτα μαζί και μετά απαντήσεις. Ρομέρο Λόπες, Γκόμες. Ε, κύριε Ρομέρο Λόπες πρώτα. Αυτός ο ιός για αυτό το malware, το κακόβουλο λογισμικό που δεν ε, μπορέσετε να μας εξηγήσετε. Γιατί, γιατί είναι τόσο εξεζητημένη τεχνολογία, τόσο περίπλοκη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τι τεχνολογία είναι. Είναι η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ε, για να ε, περάσει απαρατήρητο αυτό το λογισμικό όταν παρισέφησε τα συστήματά σας ήθελε ε, να καταστρέψει τα συστήματά σας. Ποια ήταν η πρόθεση του ιού. Απλώς θα περάσει απαρατήρητος μέσα στο σύστημα, να παραμείνει μέσα στο σύστημα απαρατήρητος και πόσο καιρό ε, λειτουργούσε έτσι το σύστημα ή μήπως ήθελε να καταστρέψει τα δικά σας συστήματα. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να πω ότι, ότι ήταν κοινικό, αγενές και αντι... Ευρωπαϊκός ο τρόπος που μας απάντησε ο εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης ότι δεν είναι θέμα ε, η Βρετανική δημόσια ασφάλεια, αλλά η Ευρωπαϊκή δημόσια ασφάλεια, η ανασφάλεια. Γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και τέτοιους, ε, τέτοιου είδους κατηγορίες για ε, κατασκοπίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Αυτή η διείσδυση, αυτή η επίθεση επηρέασε την ιδιωτική σφαίρα των ε, αξιωματούχων σας, των υπαλλήλων σας, ε, στο εσωτερικού σας ε, συστήματος ή και των πελατών σας μπόρεσε να διαβαστούν SMS μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ. Επίσης, ποιος ήταν ο στόχος αυτού του κακόβουλου λογισμικού να πολλαπλασιαστεί, να επεκταθεί, και άλλο στόχο, όπως να μεταφέρει πληροφορίες ή να εκτρέπει πληροφορίες από τα δικά σας εσωτερικά συστήματα πληροφοριών σε άλλα εσωτερικά συστήματα πληροφοριών που θα μπορούσαν, να, για παράδειγμα, να βρίσκονται στο αρχηγείο επικοινωνιών των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανικής Κυβέρνησης. Ο κύριος Κλάση, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ απαράδεκτο ότι η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκε επιδεικτικά να παραστεί στην δημόσια κρόση. Γιατί το θέμα αυτό δεν είναι μόνο δημόσια ασφάλεια ενός κράτους μέλους, αλλά εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ κοινικό να κρύβεται κανείς πίσω, πίσω από την επικουρικότητα για να αποφεύγει να λογοδοτήσει. πολύ μεγάλο τόπιμα αυτό λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα μια ερώτηση προς την Belgacom. Αυτό το επεισόδιο θα σας παροτρύνει να αναθεωρήσετε τις εσωτερικές σας διαδικασίες γιατί χρειάστηκε να προσλάβετε εξωτερικό γραφείο εμπειρογνωμόνων για να εξηγιάνετε το λογισμικό σας και να αποκαταστήσετε την ασφάλεια του δικτύου σας. Τι σημαίνει αυτό, ότι εξωτερικές εταιρείες έχουν μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη από εσά και θα συνεχίσετε αυτές τις ε, σχέσεις ε, με τις εξωτερικές εταιρείες εμπειρογνωμόνων για να μπορέσετε να έχετε πιο ταχεία ή άμεση αντίδραση στο μέλλον σε περίπτωση ανακάλυψης και νέου κακόβουλου λογισμικού. Ο κύριος Στάνταρτ. Ως προς την πρώτη ερώτηση. Ποιος ήταν ο στόχος αυτού του ιού, του κακόβουλου λογισμικού. Η υπόθεσή μας σήμερα είναι ότι ο στόχος του λογισμικού του ιού αυτού δεν ήταν να καταστρέψει το σύστημά μας. Δεν βρήκαμε ενδείξεις που να στοιχειοθετούν τέτοια πρόθεση. Άλλωστε δεν έχει επηρεαστεί η παροχή υπηρεσιών από τον ιό. Δεν έχουμε στοιχεία επίσης ότι έχει διεισδύσει, έχει ο ιός στα δεδομένα των πελατών μας. Εμείς διαπιστώσαμε την παρουσία του ιού στα τέλη Ιουνίου αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ξεκίνησε αυτή η διείσδυση, πότε ξεκίνησε αυτή η κυβερνοεπίθεση. Ακόμη δεν έχει διαλευκαθεί αυτό. Και από τεχνική άποψη είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε την ακριβή ημέρα της επίθεσης από τον ιό. Δεύτερη ερώτηση. Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Δεν βρήκαμε η κακόβουλο λογισμικό στην τράπεζα δεδομένων των πελατών μας, ούτε στο υπόλοιπο δίκτυό μας. Μόνο στο εσωτερικό σύστημα της Belgacom βρέθηκε αυτός ο ιός. Ούτε έχουμε στοιχεία που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επλήγει η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των πελατών μας. Επίσης δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα γιατί δεν έχουμε Αποδείξει για όλα αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των σχεδίων ε, ή των διαδικασιών, θα ήθελα να πω ότι η προτεραιότητα τη Belgacom είναι η ασφάλεια του συστήματο. Γι' αυτό και κάθε χρόνο, κάθε χρόνο επενδύουμε μεγάλα κονδύλια ώστε να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε την ε, τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη μας. Και χάρη στο περιστατικό αυτό βελτιώσαμε και το χρόνο αντίδρασής μας. Επαναλαμβάνω, το λογισμικό αυτό ήταν πολύ εξεζητημένο και πολύ περίπλοκο. Και πιστεύω ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την κρίση. Γιατί αντλήσαμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα και διδαχθήκαμε από τα παθήματά μας. Μάλιστα, ε, ένα πλάνο με δράση που είχαν ήδη προβλεφθεί εξαιτία αυτής της επίθεσης ε, θα εφαρμοστούν πολύ πιο γρήγορα. Σύντομη συμπληρωματική ερώτηση από την κυρία Γκόμες, αλλά πραγματικά σύντομη. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα μία απάντηση στην ερώτησή μου. Αυτό το κακόβουλο λογισμικό έδωσε τη δυνατότητα στα δεδομένα αυτά να αντιγραφούν και να μεταβιβαστούν χωρίς να καταστραφούν σε κάποιο άλλο δίκτυο πληροφορικής. Για παράδειγμα, να μεταβιβαστούν, για παράδειγμα, σε κάποιον από τις ε, Βρετανικές ε, Μυστικές Υπηρεσίες, ο οποίος θα υποκλέπτει συνομιλία κάποιων ευρωβουλευτών. Είναι ξεκάθαρη η ερώτησή σας, παρακαλώ. Ναι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποια από τα στοιχεία για να μπορούμε βασισμένοι σε αυτά να κάνουμε κάποια δήλωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ούτε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, ούτε μπορούμε να αρνηθούμε τίποτα. Έχω μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Μπιλέτ. Ο κύριος Λίτερ δυστυχώς έχει φύγει. Έχετε ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι ο δράστης είχε πρόσβαση στους δικούς σας πόρους, στο δικό σας δίκτυο, αλλά στο μέλλον δεν αποκλείεται να ξανασυμβεί αυτό και τότε είστε εκτεθειμένοι. Αναφέρετε επίσης ε, πώς πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί κανόνες και να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό είναι κάτι που θα επιληθεί σε ανώτερο επίπεδο, αλλά πώς αυτό θα μεταφερθεί στην πράξη, τι θα γίνει σε επίπεδο εταιρείας, της δικής σας εταιρείας, σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Πράγματι. Αυτό το ερώτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε ως εταιρεία είναι να διασφαλίσουμε μια επαρκή προστασία των συστημάτων μας και αυτό είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Πρέπει να δούμε ε, τα διδάγματα που θα αγγλίσουμε, πρέπει να γίνουν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με τους άλλους παρόχους. Υπάρχουν οι υποδομές, με άλλα λόγια. Επίσης, σήμερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων στην Ευρώπη, για να το θέσω έτσι, δεν είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητα. Χρειάζονται και τα αναγκαία κονδύλια, αναγκαίοι πόροι, έτσι ώστε να υπάρχει μια επαρκής και κατάλληλη πολιτική για τον κυβερνοχώρο. Και υπάρχουν πάντα περικοπές που γίνονται σε αυτούς ε, τους πόρους και αυτά τα κονδύλια. Όπως ε, σας είπα, αυτή η επίθεση δεν ήταν τυχαία. Είχε, έγινε σε μεγάλο εύρος, ήταν ε, περίπλοκη τεχνικά και είχε πίσω της μεγάλους πόρους. Ξέρω ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία στον κόσμο, καμία αρχή η οποία είναι 100% προστατευμένη από μια τέτοια επίθεση και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε ε, περιλαμβάνει συζήτηση και συνεργασία. Φυσικά και υπάρχουν μέτρα από πρόληψη μέχρι ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν. Και φυσικά αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και να δούμε ποια συγκεκριμένα μέτρα χρειάζονται και για τις εταιρείε και για τις ε, αρχές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όπως είπατε και εσείς, ε, στο ερώτημά σας αν μπορούμε να έχουμε ένα οπλοστάσιο για τέτοιες επιθέσεις, δυστυχώς οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η επίθεση έγινε σε τέτοιο επίπεδο ώστε καμία εταιρεία, καμία επιχείρηση να μην μπορεί να την αντισταθεί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό μας ε, φέρνει στο τέλος ε, της ε, συζήτησης. Να πω συμπεραίνοντας ότι αυτή η επίθεση είχε τεράστιες διαστάσεις και ο υπέτειος φαίνεται ότι ήταν κάποιος μεγάλος οργανισμός ή, κάποιος, ή κάποιο κράτος. Και ω αποτέλεσμα αυτή τη επίθεση ε, πλήγησαν μόνο τα εσωτερικά συστήματα τη Belgacom. Γιατί λοιπόν αυτό θεωρήθηκε τόσο μεγάλο και σημαντικό συμβάν ώστε να έπρεπε να αναφερθεί. Αν ήταν μόνο τα εσωτερικά συστήματα που δέχτηκαν επίθεση και κανένα τηλεφώνημα δεν υπεκλάπη, γιατί λέτε εσεί ότι πήγε η επίθεση παραπέρα από τα εσωτερικά δίκτυα τη Belgacom, γιατί να υπάρχει λοιπόν ε, στόχος μια τρίτη χώρα, όπως είπατε. Μου διαφεύγει κάπως αυτή η αιτιολογία και μπορώ να πω ότι με μπερδέψατε περισσότερο από όσο στην αρχή, πριν γίνει αυτή η συζήτηση. Όπως και να έχει όμως, ε, είμαστε ευγνώμονες που μπορέσατε να έρθετε εδώ και να μας δώσετε λεπτομερείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις μας και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις και να μπορέσουμε να σας καλέσουμε για να μας τις απαντήσετε. Τώρα ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της ε, συζήτησής μας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος, όπου ο κύριος ε, Λοβάν, όπως είπα, ο υπεύθυνος ε, της Βρετανικής κυβέρνησης έχει αρνηθεί να έρθει. Γι' αυτό λοιπόν θα περάσουμε αμέσως στον κύριο Φρανκ Ρόμπεν, τον Ευέλγο Επόπτη προστασίας δεδομένων. Την Επιτροπή δηλαδή για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του Βελγίου, όπως λέγεται εδώ, υπόπτυση προστασίας δεδομένων. Ο κύριος Ρόμπεν έχει το λόγο για μια σύντομη εισαγωγή. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να σας πω δύο τινά εκ μέρους της Επιτροπής μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Και Στη συνέχεια θα σας πω τι διδάγματα αντλήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την υπόθεση αυτή. Ο ρόλος μας εδώ στην Επιτροπή Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής είναι να δούμε αν τα μέτρα που έχουν εγκριθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αρκετά δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Και από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό αυτό, συνεργαστήκαμε αμέσως με την Belgacom που ήταν πολύ ε, πρόθυμη και μάλιστα μας ε, κοινοποίησε και τα εμπιστευτικά έγγραφα. Υπό τον όρο θα κρατούσαμε εμείς και εμείς αυτό τον απόρριτο χαρακτήρα. Αμέσως λοιπόν ενημερωθήκαμε και αμέσως ε, αντιδράσαμε για να αποφύγουμε επέκταση των ζημιών αυτής της κυβερνοεπίθεσης. Προσπαθήσαμε μέσως να μετριάσουμε τις βλάβες αυτής της διοκτήου παραβίασης. Και όπως διαπιστώσαμε δεν είχαμε διάδοση, υπονόμευση του δικτύου ή μόλυση του, των προσωπικών δεδομένων από τον ιό, ούτε μεταβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Τώρα, έχω κάποιες προτάσεις ε, να σας κάνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν να αποφύγουμε την ε, κινδυνολογία για να μην φοβίζουμε τον κόσμο. Τα, σύστημα, συστήματα πληροφορικής είναι και χρήσιμα και πολύ ασφαλή. Δεν θα πρέπει να αποτραπεί ο κόσμος από τη χρήση των ε, δικτύων πληροφορικής. Τα δίκτυα κοινωνικής τα συστήματα κοινωνική δικτύωση και το καθεξής. Υπάρχουν νομικά μέσα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων. Καλό θα ήταν όμως να αναπτύξουμε και μια πανευρωπαϊκή πολιτική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Δεν είναι θέματα που μπορούμε να αφήνουμε στις εθνικές αρχές και στα κράτη μεμονωμένα, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά όρια. Χρειάζονται υπερεθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Χρειαζόμαστε λοιπόν και νομική αντιμετώπιση, αλλά φυσικά και τη σύναψη συμφωνιών σε επίπεδο οργανισμών. Γιατί είδαμε ότι υπήρχαν κάποια μοντέλα λειτουργίας των ιών συγκεκριμένα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για τα μόντους operandi των ιών όπως είπε και ο κύριος Μπέλετ, θα πρέπει να έχουμε και ένα όγκο τεχνικών γνώσεων. Χρειαζόμαστε σημαντική τεχνογνωσία για την ανάλυση των ιών και εμείς μόνοι μας στο Βέλγιο δεν έχουμε τις αδέουσες τεχνικές γνώσεις για να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα που είναι πολύ περίπλοκα τεχνολογικά και στην ε, στο δικό μου οργανισμό έχουμε ελάχιστα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τόσο εξεζητημένες ε, και καλά οργανωμένες επιθέσεις. Δεν έχουμε καν μέσα για ε, πλήρη διαλεύκανση τέτοιων επιθέσεων. Γι' αυτό και ζήτησα μια πανευρωπαϊκή δράση. Βέβαια, όταν εκπονείται μια οδηγία ή ένα κανονισμό, καλό θα ήταν να επικεντρώνεστε τις διεθνείς πτυχές ε, και σε σημεία, σε θέματα που δεν μπορούν από μόνο τους τα κράτη-μέλη να διευθετήσουν. Καλή επικουρικότητα και θα πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά τα διασυρωριακά ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε παρευρωπαϊκό επίπεδο. Η, εγκλη... η διαμεθοριακή εγκληματικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πανευρωπαϊκά, γιατί δεν υπάρχει ένα κοινοτικό όργανο που να μπορεί να αντιμετωπίζει σήμερα τέτοιου είδους ε, επιθέσει. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και πολύ ευχαρίστω να απαντήσω στι απορίε σας. Το λόγο έχει ο εισηγητή μας για δύο λεπτά, ο Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Από ό,τι φαίνεται, δεν δίνεται σημασία στην ανάκριση για την Belgacom. Ίσως έχετε πληροφορίες. Μπορείτε να μας τις μεταφέρετε και μας για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και σε ποιο βάθος έχει πάει η έρευνα αυτή. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε επίσης και την άποψη του κυρίου Λομπάν. Δεν έχουμε τη δυνατότητα υποχρεωτική κλήτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπολογίζουμε στη συνεργασία των συναδέλφων. Οι συνάδελφοί της Belgacom μας έδωσαν τις πληροφορίες που ήθελαν σε επίπεδο συνεργασίας, αλλά ε, στη δική τους πλευρά έχουν ξεκινήσει μία νομική και ποινική διαδικασία. Δεν έχουμε τους Βρετανούς εδώ, δεν υπάρχει εκπρόσωπος λοιπόν της αρμόδιας υπηρεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας καλέσαμε όμως εσάς κύριε Ρόμπεν γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πού βρίσκονται ακριβώς οι συζητήσεις και οι ανακρίσεις. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την υπόθεση Belgacom λοιπόν και πού πηγαίνει μέχρι τώρα η ανάκριση. Εσείς μας μιλήσατε γενικότερα για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Ε, η εικόνα που μας δώσατε είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και δεν είναι σημαντική απειλή. Δεν ξέρω αν και οι συνάδελφοι κατάλαβαν το ίδιο, αλλά θα ήθελα να μου διευκρινίσετε λίγο αυτή την άποψη που εκφράσατε. Κοιτάξτε, είμαι μέλος της Επιτροπής, Ελέγχου, ε, της Επιτροπής Εγγυήσεων για την Ιδιωτικότητα. Ελέγχουμε δηλαδή το εάν τα προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων έχουν υπονομευθεί και έχουν δηλαδή χρησιμοποιηθεί για λάθος λόγους τα δεδομένα αυτά. Δεν έχουμε καμία ερευνητική εντολή για να εντοπίσουμε εμείς την πηγή ε, αυτών των διεισδύσεων. Από ό,τι γνωρίζω και θυμίζω ότι ε, έχουμε αρκετά έγγραφα από πλευρά της Belgacom στην διάθεσή μας, δεν έχουμε ε, ενδείξεις για το αν έχει υπάρξει μαζική μεταφορά δεδομένων και στοιχείων ατομικών. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή κακή αν θέλετε, ε, χρήση των δεδομένων αυτών. Πάντως η δική μας Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητες στον τομέα αυτό. Άλλες υπηρεσίες το κάνουν αυτό, όπως οι μυστικές υπηρεσίες του Βασιλείου και η εισαγγελία. Αλλά εμείς ε, ε, προσπαθούμε απλά να ελέγξουμε αν έχει υπάρξει απαράδεκτη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Κοιτάξτε, δεν ήθελα να παρανοήσω αυτά που είπατε. Σας καλέσαμε γιατί θα θέλαμε ακριβώς να μας δώσετε μια μεγαλύτερη διάσταση ανεξάρτητης ερευνητικής δραστηριότητας. Μας δώσατε μια απάντηση. Ε, η απάντηση αυτή ίσως έχει δημιουργήσει μια κάποια δυστυχία και μια κάποια απογοήτευση, τουλάχιστον να κρίνω από τον εαυτό μου. Πάντως δώσατε την απάντησή σας, ευχαριστώ δύο λεπτά. Αν κατάλαβα καλά, δεν έχει επηρεαστεί δεδομένο κάποιου πολίτη, δεν έχουν πληγεί οι πολίτες και τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο το θέμα να έχει διεθνή διάσταση, ιδιαίτερα στα πλαίσια όλων αυτών που ακούμε για το πρίσμ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια μέτρα θα, μπορούσαμε, θα μπορούσατε εσείς να λάβετε Ποιες είναι οι αιτίες και πώς έχουν πληγεί οι πολίτες. Όπως ε, είπα, εμείς είμαστε εθνικό όργανο ελέγχου, εθνική εποπτική αρχή. Και εκεί δραστηριοποιούμαστε. Πιστεύω όμως ότι είναι απόλυτα αναγκαίο, ιδιαίτερα εφόσον ε, αυτός ο ιός ήταν ιδιαίτερα τεχνολογικά περίπλοκος και δύσκολος να εντοπιστεί και να αποκρυπτογραφηθεί. Είναι πολύ σημαντικό, εάν θέλουμε να αναλυθεί αυτό από κάποιον εμπειρογνώμονα, να υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή αρχή, κάποιο ευρωπαϊκό κέντρο. Δεν μπορεί ένα κράτος μέλος, μία εθνική αρχή να λύσει το θέμα μόνη της. Μία τέτοια κυβερνοεπίθεση μπορεί να συμβεί ξανά σε, κάποια άλλη χώρα και εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες ομοιότητες. Όμως ε, το Βέλγιο από μόνο του δεν μπορεί να ερευνήσει το πρόβλημα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια κεντρική θέση και φυσικά χρειάζεται αυτή η κεντρική αρχή να είναι ικανή να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Υπάρχουν αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών και χρειάζεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε να καταφέρουμε το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα Έχουμε το σκέδιση γιατί... Θα μιλήσω εγώ σκέδιση για την Ετσάλτε. Έχοντα ακούσει τη Belgacom και τον επόπτη δεδομένων, μπερδεύομαι όλο και περισσότερο. Μιλούμε για μια μαζική, πολύ εξεζητημένη κυβερνοεπίθεση από έναν κρατικό ίσως φορέα που μια χώρα, ένας μεμονωμένος δεν θα μπορούσε να οργανώσει Βέβαια μας λέτε ότι κανένα πρόβλημα, δεν ε, μπήκαν κοργή σε τηλέφωνα, δεν έγινε μεταφορά δεδομένων, δεν έγινε υποκλοπή δεδομένων και παρόλα αυτά έχουμε μια ποινική διαδικασία που είναι απόρριτη. Πείτε μας τι συμβαίνει, το ένα ή το άλλο δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Έχουμε πραγματικά ένα ε, περιστατικό μεγάλων διαστάσεων, μια μαζική κυβερνοεπίθεση που δικαιολογεί μια ποινική διαδικασία και την σημερινή δημόσια κρόση και την διεξαγωγή έρευνων ή πρόκειται για ένα ασήμαντο περιστατικό εντός της Υπεργακόμ. Δεν μπορεί και τα δύο να ισχύουν. Δεν μπορεί να είναι από κύμα της φαντασίας το μέσο και ενημέρωσης όλα αυτά. Δεν μπορεί να τα επινόησαν όλα οι εφημερίδες. Ούτε να μας λέτε εσείς ότι ήταν υπερβολικά όλα αυτά και δεν υπάρχει πρόβλημα με καμία κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι η, ο, ο Βέργος δεδομένων δεν, μπορεί να, δεν έχει τις αρμοδιότητες να κάνει την, την έρευνα. Αλλά δεν αρκεί να λέτε ότι αρκεί κοινοτική νομοθεσία για να ε, βελτιωθούν τα συστήματα. Πρόκει, ε, για μαζική κυβερνοεπίθεση ή όχι. Γιατί αν δεν ήταν μαζική, τότε να κατεβάσουμε τα ρολά και να πάμε για μια μπύρα. Αλλιώ, αν ήταν όντω μαζική, χρεια... χρειαζόμαστε κάποιε απαντήσει. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Μέχρι στιγμής και πριν την επίθεση αυτή, ε, η Βελγακόμ απέκρο οποιοδήποτε ε, ιούς ε, προηγούμενους και κυβερνοεπιθέσεις. Πρώτη φορά βρήκαμε τέτοιο επικίνδυνο και κακόβουλο λογισμικό που ε, χτύπησε πάνω από 120 συστήματα του εσωτερικού μας δικτύου. Και αυτό δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, ε, μερικές φορές ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φουσκώνουν τα πράγματα και λένε πολλά και διάφορα, αλλά στηρίζονται σε οικοτολογίες. Εμείς ξεκινάμε από αριθμητικά στοιχεία, από πραγματικά περιστατικά και μέχρι στιγμής ε, τα στοιχεία δεν μας ε, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έγινε μεταφορά δεδομένων ε, των πελατών μας προς το, το σύστημα του δράστη της κυβερνοεπίθεσης. Και φυσικά συνεχίζουμε τις έρευνες με τις αρμόδιες αρχές και όπως είπε και ο Ντύρκ έχουμε πλήρη συνεργασία, στη συνεργασία με την Βελγική Επιτροπή Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε στα πραγματικά περιστατικά. Όντως ήταν σοβαρή η επίθεση, σοβαρή η διείσδυση που έβαλε κατά της ακαιρεότητας ε, του συστήματος και είναι η πρώτη φορά που είχαμε τόσο επικίνδυνο ιό στο σύστημα πληροφορικής. Ήταν πολύ σοβαρή κατάσταση για μας ο κύριος Ρόμπεν. Φυσικά ήταν σοβαρή κατάσταση, φυσικά ήταν σοβαρή επίθεση, αλλά ελήθησαν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και μετριάστηκαν οι ζημίες. Σίγουρα δεν υπήρχε διαρροή δεδομένων. Μία συμπληρωματική ερώτηση. τότε τι υπάρχει στο εσωτερικό σύστημα της Belgacom, στη εσωτερική διοίκηση της Belgacom που είναι τόσο ενδιαφέρον και δελαστικό ή ελκυστικό για μυστικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας ή οποιοδήποτε άλλο κράτους. Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις, αλλά δεν είναι αυτός ο δικός μου ρόλος, να κάνω υποθέσεις. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σήμερα, καμία απόδειξη και δεν ξέρουμε σε τελική ανάλυση ποιο ήταν ο στόχο αυτή τη κυβερνοεπίθεση. Ούτε καν αυτό δεν γνωρίζουμε. Ο κύριο Ρόμπεν ουδέν σχόλιο επιπλέον. Μάλιστα. Ο κύριος Άλμπρεχτ από του Πράσινου. Um, Ευχαριστώ για τον κύριο Ρόμπεν. Έχω μία μικρή σύγχυση σε σχέση με αυτό που μας είπατε Είπατε ότι όλα είναι καλά, όλα είναι τέλεια, ενώ βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσης σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ακόμα και στο Βέλγιο και το γνωρίζετε. Ξέρετε ότι παραβιάζεται και αγνοείται ο βελγικός νόμος και οι βελγικές ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και σαν μέλος της Επιτροπής Προστασίας της Ιδιωτικότητας θα έπρεπε να είσαστε λίγο περισσότερο απασχολημένος και ανήσυχος. Ελπίζω αυτό που μας είπατε να μην είναι γενικότερα η άποψη της Επιτροπής σας. Μιλήσατε επίσης και για μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ανακριτικών διαδικασιών, ερευνητικών διαδικασιών κτλ. Οι βελγικές αρχές και η βελγική αρχή έχει χρησιμοποιήσει την EC3, δηλαδή την υπηρεσία της Europol που ασχολείται με το κυβερνοέγκλημα και ζήτησε την βοήθειά της. Γι' αυτό την δημιουργήσαμε την EC3. Έχουμε εξοδέψει εκατομμύρια για να το κάνουμε αυτό. Οι βελγικές αρχές λοιπόν ζήτησαν τη βοήθεια της Europol και γιατί αν δεν το έκαναν, γιατί δεν το έκαναν. Ο κύριος Ρόμπεν. Νομίζω ότι εμείς παίξαμε πλήρως τον ρόλο μας. Σας είπα ποιος είναι ο ρόλος μας σαν Επιτροπής Προστασίας της Ιδιωτικότητας εμείς ε, ελέγχουμε την πιθανή επιμόλυνση των ιδιωτικών δεδομένων. Από ό,τι φαίνεται, ε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, με όλους τους ελέγχους εσωτερικούς, εξωτερικούς, εμπιστευτικούς, δεν έχει υπάρξει τέτοια υπονόμευση και επιμόλυνση των προσωπικών δεδομένων. Τώρα, πέρα από αυτό υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναζητεί τον δράστη. Τι έχει επίσης ε, τι έχει επιμολυνθεί, τι έχει ε, χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά κτλ. Γι' αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει εμπειρογνωμοσύνη και βελγική και ε, διεθνή. Αλλά σας είπα, εμείς δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Αυτό το κάνει η Belgacom και οι επίσημες ε, κυβερνητικές υπηρεσίες. Εμείς απλά ελέγξαμε την ποιότητα των ατομικών και προσωπικών δεδομένων και θεωρούμε ότι τα μέτρα που έλαβε η Belgacom για να προστατεύσει το σύστημα είναι τα κατάλληλα. Το ότι ελήφθησαν αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα είναι σαφές αλλά τα μέτρα είναι σωστά και αυτό θα έχει ε, σαν συνέπεια τέτοια ατομικά δεδομένα, εμπορικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα να μην επιμολύνονται. Συμπληρωματική ο κύριος Άλμπρεχτ. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι πώς μπορεί κανείς να αποκλείσει στην συγκεκριμένη περίπτωση τα ατομικά στοιχεία και δεδομένα δεν έχουν θυγεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, δεν με αφήνει ήσυχο. Έχετε κάποιες ενδείξεις, έχετε αποδείξεις ότι δεν έχουν φυγεί τα ατομικά δεδομένα. Ή δεν γνωρίζετε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία μπορεί να έχουν φυγεί. Δεν μπορώ να το αποκλείσω κύριε Άλμπεχτ. γιατί τα δεδομένα τα οποία έχουν μεταφερθεί έχουν μεταφερθεί με κρυπτογραφικό τρόπο και με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπορούμε εμείς να αποκρυπτογραφήσουμε. Αλλά ε, σε σχέση με τον όγκο, την ποσότητα των δεδομένων δεν έχει υπάρξει μαζική μεταφορά. Για το ποια είναι τα δεδομένα αυτά τότε θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουμε τον, ε, τον δούριο ύπο αν θέλετε. Θα πρέπει να σπάσουμε τον κώδικα του συγκεκριμένου κακόβουλου λογισμικού και δεν έχουμε εμείς τις αρμοδιότητες αυτές. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την αποκρυπτογράφηση. Αν είχαμε την αποκρυπτογράφηση δεν θα, ήμασταν πιο σίγουροι, αλλά σε επίπεδο ποσοτικό δεν έχει υπάρξει μαζική μεταφορά δεδομένων. Από τον όγκο των μεταφερθέντων δεδομένων ε, δεν έχει υπάρξει πρόβλημα. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε 100% ότι δεν έχουν μεταφερθεί, μεταφερθεί δεδομένα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. 100% δεν μπορώ να σας το πω. Λοιπόν, η, ομάδα των συντηρητικών ε, είναι απούσα. Έχει το λόγο η κυρία Έρντ. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε και οι δύο πριν ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί να προστατευτεί από μόνη της ατομικά. Από την άλλη, Είπατε εσείς ο επόπτης δεδομένων ότι τα κράτη έχουν ε, λίγες δυνατότητες να διερευνήσουν από μόνα τους σε τι έχει συμβεί και ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή αρχή. Θα σας ρωτήσω ευθέω. Δεν υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή καμία τεχνολογία η οποία να μπορεί να αποτρέψει τέτοιες ε, σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις. Πόσο ασφαλής είναι η Belgacom πρώτον πόσο ασφαλής είναι η ιδιωτική ζωή των πολιτών. Τεχνικά μιλώντας μόνο, πρώτον και δεύτερον. Θα αρχίσω από την άλλη αυτή τη φορά. Και τι έρευνες έχουν γίνει σχετικά με την ασφάλεια και την Belgacom, ποιοι έλεγχοι έχουν διεξαχθεί, σε ποια διαστήματα, ποια ήταν τα αποτελέσματα, πότε ήταν ο τελευταίος έλεγχος και ποιος κάνει αυτούς τους ελέγχους. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι κάτι άλλο. Και τι θέλετε να κάνετε σε σχέση με την αποκρυπτογράφηση, τι θέλετε να αλλάξετε στο μέλλον. Και τώρα όσον αφορά το... αυτά που διάβασα στο Spiegel για, ε, για αυτό που έγινε. Εσείς λέτε ότι τα εσωτερικά συστήματα μόνο επλήγησαν. Ωραία. Τα εσωτερικά συστήματα που επλήγησαν θα πρέπει να είχαν χειριστεί από ανθρώπους, δεδομένα των οποίων θα υπήρχαν σε αυτά τα συστήματα. Ε, αυτοί τι έγιναν. Νομίζω ότι για τα πραγματικά περιστατικά αρμόδια είναι να απαντήσει η Βελγακόμ. Αν ήταν δυνατόν να αποφευθεί η κυβερνοεπίθεση, δυστυχώς ε, μάλλον όχι. Γιατί από τη στιγμή που ένας ιός μπορεί να μπει από μεταθύρες στο σύστημα, είναι πολύ δύσκολο το σύστημα να τον αποκρούσει. Στις Ηνωμένε Πολιτείες μα είπαν ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα στεγανό και αδιάβλητο. Για να έχουμε απόλυτα αδιάβλητα και στεγανά συστήματα θα πρέπει να τα ελέγχουμε διαρκώς και παγκοσμίω. Δεν αποκλείεται λοιπόν όταν αγοράζουμε λογισμικό από μια εξωτερική επιχείρηση ότι δεν θα υπάρχει μια κρυφή πόρτα στο σύστημα. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λάβουμε μέτρα δεδομένου του κινδύνου και της προηγμένης τεχνολογίας, του κόστους και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού τους κινδύνους, αλλά να τους αποκλείσουμε πλήρως αποκλείεται ο εκπρόσωπος της Belgacom. Θα ήθελα να πω ότι η αποκατάσταση ασφάλειας του συστήματος πληροφορικής για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε ε, να επεξεργαζόμαστε μέτρα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια και να προλάβουμε μελλοντικές ε, παραβιάσεις του δικτύου μας. Είχαμε και στο παρελθόν μια κυβερνοεπίθεση που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αν είχαμε τα σημερινά μέτρα. Σε ό,τι αφορά του τεχνικούς κανόνες, εφαρμόζουμε τις υψηλότερες διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές. Και το σύνολο των δεδομένων μας έχει το πρότυπο ίσο. Οι προδιαγραφές μας λοιπόν είναι πολύ αυστηρές και ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγχτές. Επίσης έχουμε και γνώμονες ε, και συγκριτικά μέτρα για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις δικές μας επιδόσεις με άλλους ε, αντίστοιχους ε, παρόχους. Συμμετέχουμε και σε μια επιτροπή δεοντολογίας. Βέβαια, όταν μιλούμε για ασφάλεια, δεν μιλούμε μόνο για αρχιτεκτονική του συστήματος, αλλά και δράσεις σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και για μια κουλτούρα ασφάλειας σε μια επιχείρηση. Και μάλιστα αυτά τα benchmark που έχουμε, ε, κανόνες σύγκρισης, μας οδηγούν σε συμπεράσματα, αντλούμε κάποια διδάγματα και κάθε χρόνο ε, επικαιροποιούμε και ενισχύουμε τα μέτρα ασφάλειάς μας. Έχουμε αφενός την εσωτερική μας υποδομή του συστήματος πληροφορικής, αλλά και εξωτερική υποδομή. Άιλη, που παρέχουμε στους ε, πελάτες. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ε, ο αδύναμος κρίκος στο εσωτερικό μας σύστημα και από πού μπήκε αυτός ο ιός. Τώρα, αν θα αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας ε, ή αν το αλλάξαμε. Ναι, έχουμε ενισχύσει τον τρόπο λειτουργίας μας, έχουμε εγκρίνει συμπληρωματικά μέτρα, έχουμε εντατικοποιήσει το monitoring, την παρακολούθηση που κάνουμε και μάλιστα αυτή τη στιγμή εκπονούμε και τεχνικό έλεγχο. Η σχετική έκθεση θα υποβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πελγακόμ, ώστε να αντιλήσουμε τα συμπεράσματα από την κρίση αυτή και να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας για το μέλλον. Για να ολοκληρώσουμε με τους κοιόδης ηγητές, η κυρία Μορβάη από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Προστασίας της Ιδιωτικότητας για την παρουσία του. Ίσως να παρανόησα αυτό που είπατε και θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε. Μας είπατε ότι από τη μία είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μία μείζον κυβερνοεπίθεση στην Belgacom. Από την άλλη είπατε ότι δεν έγινε ιδιαίτερη ζημία στους πελάτες, οπότε το θέμα δεν σας αφορά ακριβώς και δεν θα ασχοληθείτε με αυτό. Και σκεφτόμουν παράλληλα ότι αν κάποιος πυροβολεί προς την κατεύθυνση κάποιου και η σφαίρα δεν τον πετύχει, τότε σε αυτή την περίπτωση η, αστυνομία θα πει εντάξει σκοτιστήκαμε και που έγινε πυροβολισμός δεν χτύπησε κανένα Οπότε θα πρέπει ίσως να προστατεύεται καλύτερα μόνο του το θύμα από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να, υπα... να θεωρηθεί σαν απόπειρα φόνου, συνεπώς ποινικά κολάσιμη. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωση. Και από ό,τι φαίνεται επίσης οι βελγικές αρχές, ιδιαίτερα η εισαγγελία, ε, χρειάζεται βοήθεια στα πλαίσια αυτής της έρευνας και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και είναι σε θέση ίσως να βοηθήσουν. Ε, υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ακούσαμε την άποψη της εισαγγελία για λόγους που δεν γνωρίζουμε. Είναι ότι ο Έντουαρντ Σνόου, ο Σνόουντεν γνωρίζει πολλά για αυτή την περίπτωση, έστω και μέσω του Skype. Θα μαγνητοφωνήσουμε αυτά που θα μας πει και θα τα υποβάλουμε στην Βελγική Εισαγγελία σαν υλικό το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οπότε η κατάσταση θα γίνει ξαφνικά πολύ πιο εύκολη γιατί είναι ε, χρήσιμο γενικά να το κάνουμε. Εξαιρετική ε, Συμβουλή σίγουρα η Belgacom θα μας παράσχει μια σύνδεση ασφαλέστατη με το Skype. Κοιτάξτε, ε, να το διευκρινίσουμε. Έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής εξετάζονται τα γεγονότα τα οποία πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις, για τα οποία πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Μέσα σε όλα αυτά είναι και η δική μου επιτροπή η οποία δεν έχει ούτε ερευνητικέ διαδικασίες ούτε ποινικέ διαδικασίες ω εκ τούτου δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Τώρα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα εμείς ελέγξαμε αν κάποιες ενέργειες που έγιναν είναι αντίθετες με την ενισχύη νομοθεσία και είδαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων. Ε, ε, εμείς εκεί σταματάμε σαν Επιτροπή Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Ελέγχουμε αν υπονομεύθησαν τα προσωπικά στοιχεία, τα ατομικά στοιχεία των Βέλγων πολιτών, των πολιτών γενικά. Δεν έχει διαπιστωθεί μια τέτοια παραβίαση. Ελέγξαμε επίσης αν τα μέτρα που έλαβε η Μπελγκακόμ είναι επαρκή για να αποφευθούν τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον. Είναι. Και τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία η αντίδραση της Belgacom ήταν η κατάλληλη, φυσικά και ήταν, οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα εισαγγελία. Τα δικαστήρια στο Βέλγιο θα ασχοληθούν με τα υπόλοιπα δεν έχετε προσκαλέσει εκπρόσωπο της δικαιοσύνης, έχετε προσκαλέσει ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα έπρεπε να προσταλέσετε ανθρώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο εγώ. Ή κάποιον που να ε, αντιπροσωπεύει το ποινικό κομμάτι, εν περιπτώσει, που να ασχολείται με την δίωξη ε, εις βάρος τέτοιου είδους ενεργειών, σε ποινικό επίπεδο. Λοιπόν, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Έχουμε ε, ε, μελέτες, έχουμε έρευνες οι οποίες συνεχίζονται. Μια διευκρίνηση. Θεωρείτε ότι το σημαντική περίπτωση παραβίασης της ιδιωτικότητας. Παρόλο που μπορεί να μην ε, υπήρχε πρόσβαση στα δεδομένα των ε, ατόμων υπήρξε κίνδυνος όμως τέτοια παραβίασης. Δεν ξέρω τι κανόνες διέπουν το έργο της Επιτροπής σας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είστε αρμόδιος για τα θέματα αυτά. η Επιτροπή σας προστατεύει την ιδιωτικότητα, την ιδιωτική σφαίρα των ε, κατοίκων του Βελγίου, υπήρξε πολύ σοβαρός κίνδυνος ε, παραβίασης της ιδιωτικής σφαίρας, οπότε θεωρώ ότι και είστε αρμόδιοι στην περίπτωση αυτή η επιτροπή σας δηλαδή. Καλά, δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση. Ο κύριος Ρόμπεν, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, ήταν σοβαρή η επίθεση και θα πρέπει να αποκατασταθεί η ασφάλεια του συστήματος. Σε ό,τι αφορά την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, στο θέμα αυτό δεν είχαμε παραβίαση τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας. Προβλήματα ασφάλειας, ναι, υπήρξαν σοβαρά και θα πρέπει να ρυθμιστούν. Αλλά δεν υπήρξε διαρροή προσωπικών δεδομένων των πελατών της Belgacom. Οπότε δεν αμφισβητήθηκε ή δεν επλήγει η ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας που έχει μια συμπληρωματική ερώτηση, μια σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Ρόμπεν. Καταρχήν ε, αντιλαμβανόμαστε τους περιορισμούς ε, της Επιτροπής σας, μια και έχει ξεκινήσει και δικαστική έρευνα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας ε, άλλα στοιχεία της βελικής υποδομής ή δικαστικής που έχουν υπο... πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Γιατί σε, σε συνεργασία με την Europol έχουμε αυτό το κέντρο ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ακριβώ για να αποφύγουμε τέτοιε κρίσει και περιπτώσει. Αλλά κανένα κράτο ε, δεν έχει πρόσβαση σε αυτή την υποδομή. Κανένα δεν τη χρησιμοποιεί. Ενώ έχουμε ένα κοινό παρανομαστή εδώ. Γιατί να μην αξιοποιείται. Αντιλαμβάνεστε ποιες είναι οι υποδομές ε, στο Βέλγιο δεν σας καλέσαμε εδώ για να σας υποχρεώσουμε συνεργασία, αλλά θα ήθελα να μας ε, πείτε αν υπάρχει κανείς που επιθυμεί ή που έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και αν ε, δεν το χρησιμοποιούν επαρκώς οι ενδιαφερόμενοι, γιατί. Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ για εκ μέρους των ε, αρχών ασφάλειας, των υπηρεσιών ασφάλειας του Βελγίου. φαντάζομαι ότι οι αρμόδιες αρχές ήρθαν σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αλλά εγώ δεν το γνωρίζω. Πάντως, αν μιλούμε για ευρωπαϊκές ε, αρμοδιότητες, θα πρέπει, αν υπάρχουν, να τις αξιοποιούμε. Ο κύριος Άλμπρεχτ, διαδικαστικό. Ε, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να σημειωθεί ότι μόλις τώρα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν κάποια αρχεία, επιβεβαιώθηκε αυτό από δημοσιογράφους, ότι υπάρχουν κάποια αρχεία τα οποία μεταβιβάστηκαν στις ε, βρετανικές ε, μυστικές ε, υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε αυτό. Εάν όμως αληθεύει, τότε αναμένω πιο ευθείε απαντήσει από πλευρά βελγικών αρχών. Ε, η πρόεδρο ε, ζητάτε επαλήθευση από ποιον ακριβώ, από την Belgacom ή από τον επόπτη προσωπικών δεδομένων. Εσεί θα μου απαντήσετε όποιο θέλει, αλλά είναι απογοητευτική η έλλειψη επιβεβαίωση και να μαθαίνουμε κάτι τέτοιο από δημοσιογράφου. Ωραία, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν και του δύο και την Μπέλγα ακόμα και τον επόπτη προστασία δεδομένων να απαντήσουν και θα περάσουμε στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Εάν αληθεύει αυτό που ισχυρίζονται οι δημοσιογράφοι, τότε πράγματι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι λαμβάνουμε τις πληροφορίες μετά από αυτούς. Ε, δεν έχουμε όμως εμείς προς το παρόν κάποιες ενδείξεις σχετικά με το ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση. Ο κύριος Ρόμπεν, δεν έχω κάτι να προσθέσω, δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Μάλιστα. Η κυρία Σίπελ, η κυρία Γκόμες, η κυρία Ρομερο τώρα θα λάβουν το λόγο, η κάθε μία για μισή λεπτό και έπειτα θα επιστρέψουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ήταν πολύ περίεργη η τελευταία συζήτηση, το τελευταίο πάνελ. Πολλές φορές ε, ακούσαμε σήμερα για αυτήν την επίθεση και για αυτά τα κονδύλια που χρειάζονται, αυτοί, αυτούς τους πόρους που χρειάζονται, την οργάνωση. Και ακούσαμε επίσης ότι ε, καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν έχει αυτούς τους πόρους ε, στη διάθεσή της. Ποιος όμως θα μπορούσε, αν όχι μια μυστική υπηρεσία. Δεύτερον, εάν όντως ήταν μια μυστική υπηρεσία πίσω από αυτή την επίθεση και όχι κάποια εταιρεία τότε. Αυτό αποτελεί παρασβίαση πολλών ε, νόμων ευρωπαϊκών, αλλά ρωτώ ποιος έχει τις τεχνικές δυνατότητες αποτροπής μιας τέτοιας επίθεσης. Αν όχι μυστικές υπηρεσίες. Τρίτον, μας λέτε ότι δεν επλήγησαν προσωπικά δεδομένα πελατών, ότι δεν έγινε επίθεση και από την άλλη. Αναφέρεστε στο ότι χτυπήθηκε το εσωτερικό δίκτυο της Belgacom. Όμως αυτή η επίθεση δεν έχει δεν είχε στόχο τους πολίτες, τους πελάτες. Αυτός δεν ήταν ο τελικός στόχος. Κυρία Γκόμες. Κύριε Ρόμπεν, είπατε ότι δεν έχετε αποδείξεις για μαζική μεταφορά δεδομένων. Έχετε μήπως στοιχεία για μια επιλεκτική μεταφορά, αντιγραφή ή περί τυχαία παρακολούθηση κάποιων μηνυμάτων έστω και προσωπικών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση. Δεν μιλούμε για μαζική μεταφορά, έστω και επιλεκτική ή τυχαία ή επιλεκτική παρακολούθηση. Κανένας δεν περιμένει ε, έρευνες από την Europol φαίνεται και το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Γιατί να μην αποταθούμε εμείς σε αυτό το κέντρο ασφάλεια στον κύριο Δεν έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε εμείς να λάβει δράση. Δεν είστε δυστυχώς κράτος κυρία Γκόμες. Δεν δικαιούστε να προσφύγετε. κυρία Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή μας μιλήσαμε πολλάκι για την ε, δυνατότητα των εργαστηρίων για κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δεδομένων. Στο Βέλγιο, τι εργαστήρια ασχολούνται με τέτοια κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δεδομένων. Ε, τα εργαστήρια αυτά, οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν τόσο τεράστια ευθύνη θα πρέπει να είναι γνωστές και επίσης να λαμβάνουν συγκεκριμένη πιστοποίηση και αδειοδότηση για να ξέρουμε αν όντως ανταπεξέρχονται στο ύψος των ευθυνών τους και των περιστάσεων και να ξέρουμε και πώς λειτουργούν γιατί είναι οι ίδιες επιχειρήσεις, τα ίδια εργαστήρια που χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί, θα πρέπει τέτοια στοιχεία να είναι στη διάθεσή μας. Μάλιστα, τρεις ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρόμπεν για να απαντήσει και μετά στους εκπροσώπους της Μπέλγα αν το επιθυμών. Θα είμαι σύντομος. Θα για την αποκρυπτογράφηση, την κωδικοποίηση αν θέλετε. Αποκωδικοποίηση. Οι πληροφορίες που ξέφυγαν από το σύστημα, βγήκαν από το σύστημα, ήταν κωδικοποιημένες όχι από την Belgacom, αλλά ο ιός που χρησιμοποιήθηκε εμπεριέχει κρυπτογραφικές τεχνικές για να αποκρύβει τα στοιχεία τα οποία υφαρπάζει Συνεπώς θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε πρώτα τον ιό και μετά να μιλήσουμε για πιθανή ε, ε, ανάγνωση των, στοιχείων που μεταφέρθηκαν. Για να δούμε το περιεχόμενο των στοιχείων που διέφυγαν θα πρέπει να έχουμε περάσει στην αποκωδικοποίηση. Δεν είναι λοιπόν το γεγονός ε, ότι η αποκωδικοποίηση κρυπτογράφησε τα δικά της δεδομένα. Όχι, ο ιός είναι αυτός ο οποίος κωδικοποίησε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορούμε εμείς να αναγνώσουμε την ποιότητά τους. Το τι ακριβώς ε, έχει υπάρξει σε επίπεδο λεπτομέρειας ε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, η ανάκριση θα το δείξει, θα δούμε ποιο είναι το επίπεδο επιμόλυνσης. Ίσως να υπήρξαν επιλεκτικές μεταφορές, ίσως διευθύνσεις ηλεκτρονικές ταχυδρομείου. Δεν το ξέρουμε όμως. Πάντως δεν έχει υπάρξει μεγάλος όγκος δεδομένων που έχει μεταφερθεί. Η Μπελγκακόμ έχει το λόγο. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις για μεταφορά στοιχείων των ε, πελατών μας. Φυσικά και γνωρίζουμε ότι έχουν διαφύγει μέσα από τις λεγόμενες μεταπύλες ε, κάποια ε, στοιχεία τα, η υπόλοιπη διαδικασία, η ανακριτική, νομίζω ότι θα διευκρινίσει ακριβώς ε, το τι έχει γίνει. Τώρα το ποιος είναι ο δράστης. Είναι μια μυστική υπηρεσία άλλης χώρας ή όχι. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα τέτοιο λογισμικό έχει τα μέσα. Ποιος κρύβεται πίσω από το λογισμικό αυτό μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουμε. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε η Βρετανική Αρμόδια Υπηρεσία να σας βοηθήσει να τα αποκρυπτογραφήσετε. Η κυρία Μόρθο ε, διαδικαστικό. Είναι πραγματικό ή πολιτικό. Έχετε πρόβλημα με την πολιτική. Νόμιζα ότι είσαστε πολιτικός και εσείς και εγώ. Πιστεύουμε και οι δύο στην πολιτική. Για το διαδικαστικό του κυρίου Άλμπρεχτ. Από ό,τι φαίνεται ότι ό,τι στοιχεία, ό,τι αποδείξεις έχουν συλλέξει μάρτυρες και δημοσιογράφοι αντιμετωπίζονται σαν φήμες Ας δημιουργήσουμε λοιπόν ένα χώρο, ένα πλαίσιο έτσι ώστε να μετατρέψουμε τις φήμες σε αποδείξεις. Σας είπα το παράδειγμα του Σνόουντεν. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με όλες τις επιφυλάξεις γύρω από την περίπτωση της Belgacom και με, να τα μεταφέρουμε στην εισαγγελία. Δεν ξεπερνούμε έτσι τις αρμοδιότητές μας αλλά βοηθάμε τις ποινικέ διαδικασίες. Μην ανησυχείτε ότι αν έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία θα τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις ε, κύριε εισηγητά. Κοιτάξτε, όταν κλείσει η έρευνα θα υπάρξουν και τα τελικά συμπεράσματα. Προς το παρόν θέλω να ευχαριστήσω τους μάρτυρες που ήρθαν εδώ. Δεν ε, κλήθησαν, όπως είπα, υποχρεωτικά. Ήρθαν επειδή επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας. Όπως είπαμε ακριβώς έχουμε μια περίπτωση prima face. Ε, κινήθηκε κατά συνέπεια η Βελγική εισαγγελία και γι' αυτό εμείς δεν έχουμε προχωρήσει σε σχέση με το ποιους ξεκίνησαν τη διαδικασία, ε, υποθέσεις κάνουμε, αλλά εμείς σαν πολιτικοί δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουμε σε επίπεδο αν θέλετε ενημέρωσης, ε, ε, μας λείπουν τα στοιχεία που δεν μας μετέφερε η Βρετανική πλευρά, ε, δεν έχουμε μια πλήρη ανεξάρτητη ανάλυση από πλευρά των βελγικών αρχών, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένες υποθέσεις. Σαν παράδειγμα ότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το κέντρο δίωξης κυβερνοεγκλήματος, αυτό είναι αρκετά σαφές δεν θα κλείσω λοιπόν με επίσημα συμπεράσματα, νομίζω όμως ότι η συνάντηση ήταν μια χρήσιμη συνάντηση γιατί πράγματι θέσαμε πολλές έγκυρες ερωτήσεις, πήραμε κάποιες ε, σαφείς ε, και κάποιες λεγότερο σαφείς ε, απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά. Να σας ευχαριστήσω όλους όσους ήσασταν εδώ πέμπτη απόγευμα και θέσατε τις ερωτήσεις σας και όσους μας παρακολούθησαν στο διαδίκτυο. Και εγώ λέει η Πρόεδρος Ιντβέλτ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Σας κάναμε τη ζωή δύσκολη, δεν ήταν προσωπικό όμως αυτό. Νομίζω ότι όλοι φεύγουμε από τη συνάντηση αυτή με περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Δεν φταίτε εσείς γι' αυτό ίσως, αλλά δεν έχετε πλήρης ανακριτικές διαδικασίες. Δεν έχουμε κι εμείς ε, την ε, δυνατότητα επιβολής ένορκης μαρτυρίας <clears throat> αλλά εφόσον και το Βελγικό Κοινοβούλιο κάνει μια τέτοια ε, ακρόαση θα ζητήσει να καταθέσετε μετά από ορκομοσία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ε, θα δοθούν απαντήσεις σε κάποια θέματα γιατί όπως είπατε δεν ξέρουμε το μέγεθος, δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, δεν ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο οπότε όλες οι αναφορές του τύπου είναι στον αέρα πια, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Η επόμενη λοιπόν συνάντηση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 7 ε, το απόγευμα στο Στρασβούργο.